ο οποίος ε, έμεινε εδώ μέχρι το τέλος της συζήτησης. Η συνεδρίαση συνεχίζεται αύριο στις 26 Οκτωβρίου από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 και 11.30 με 1.30. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και ε, μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καληνύχτα σε όλους και ευχαριστώ τους Ιρμήνους και πρόεδρους.